Συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην απογευματινή συνεδρίαση. Περνάμε στο σημείο υπαριθμών 9, πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία, που αφορά σχέδιο γνωμοδότησης για τη σύνοση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο Πέτρας Αουστρεβίτσιο. Θέλετε το λόγο, κύριε Σιγητά. Όχι. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. One vote Okay, no, one, Εγκρίνεται με 57 υπέρ 3 κατά ψήφους. Περνάμε στο σημείο 10. Γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη Σύμβαση Συμφωνία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λευκορωσία για την επενδυσδοχή προσώπων που διαμένουν χωρί άδεια για άλλη μια φορά. Συντάξει γνωμοδότηση είναι ο κύριος Αστρεβίτσιος, θέλετε το λόγο. Όχι, απογοητευόμαστε όλοι. Δεν πειράζει, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται και αυτή με 53 ψήφους υπέρ 10 κατά. Και περνάμε στο σημείο 11. Σύσταση προς τον ύπατο εκπρόσωπο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 118, για την προετοιμασία της διαδικασίας επανεξέτασης της συνθήκης περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις δυνατότητες πυρηνικού αφοπλισμού. Η συγκητής είναι ο Σβεν Μίξερ. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι τόσο ταπεινός όσο ο συνάδελφος Πέτρας, οπότε εγώ θα τοποθετηθώ. Ε, φέτος η φετινή συνδιάσκεψη αποτελεί την 50η επέτειο της θέσης ισχύ της ε, συνθήκης όμικρον, ε, σίγμα μη δέλτα που αποτελεί το πλαίσιο για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη διευκόλυνση της χρήσης μη στρατιωτικής ε, χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της εξάπλωσης των ε, πυρηνικών όπλων και είναι προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση το γεγονό ότι στέφτηκε η φετινή συνδιάσκεψη με επιτυχία, όχι μόνο γιατί αποτέλεσε την ε, επέτειο τη συνθήκη αυτή, αλλά γιατί και η αποτυχία επίτευξη συμφωνία όσον αφορά το τελικό έγγραφο θα αποτελούσε τη δεύτερη στη σειρά αποτυχία καθώς πριν από πέντε χρόνια υπήρξε μια σχετική διάσκεψη η οποία δεν κατάφερε να καταλήξει σε ένα έγγραφο συνένεσης. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που δραστηριοποιήθηκαν ενεργότατα, που συμμετείχαν στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου μέσα από μεγάλο αριθμό τροπολογιών, πολλές εκ των οποίων θεωρώ ότι αποσαφηνίζουν και ενισχύουν την αρχική στήσταση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδίως τους σκιώδους, σκιώδεις εισηγητές με τους οποίους είχαμε επικοδομητικές συζητήσεις και με τους οποίους καταφέραμε να συντάξουμε και να συνδιαμορφώσουμε 10 συμβιβαστικές τροπολογίες στη βάση όλων των τροπολογιών που είχαν κατευθεί και ελπίζω να τύχει η έκθεση αυτή της υποστήριξης τόσο της Επιτροπής ΑΦΕΤ όσο και της Ολομέλεια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν δεν θα ήθελε κάποιος άλλος να τοποθετηθεί, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ με τις κάρτες σας, επί της τροπολογίας 50. Πέρας της ψηφοφορίας Μάλιστα. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ επί της τροπολογίας 53 πέρας απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να το ελέγξουμε να είμαστε σίγουροι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 54. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Ψηφίστε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 56. Πέρας. Εγκρίνεται και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. 57 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Επί 66 η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να το ελέγξουμε γιατί δεν ήταν πολύ εμφανές. Ψηφίστε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Παρακαλώ, ας το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. It's closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά κιόλας. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 73 κατά πίπτη. 74. Όχι, δεν εγκρίθηκε 71. Οπότε ψηφίζουμε επί της 74. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό. Ψηφίστε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 απεσύρθη, 87 υπέρ, κατά αποχές δεν ήταν πολύ σαφές, οπότε καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά επί 87. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Επαληθεύουμε μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίστε σας παρακαλώ επί της 91. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά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 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε καλύτερα για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 113 του κυρίου Ντανζόν. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 δεν έχει ληφθεί υπόψη. 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ετυλογικές σκέψεις 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε επί της 7 ε, πέρας της οφορίας. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει και περνάμε Στη 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της 16 γιατί ζητήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εμένα μου φάνηκε πολύ σαφές το αποτέλεσμα, αλλά δεν πειράζει. Α το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Ε, ναι. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά Αποχέ. θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και με μεγάλη διαφορά. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές, θα το ελέγξουμε. Ψηφίστε σα παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της 20. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 που την έχει υιοθετήσει ο Πέτρας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης ή ε, ακούσιας χρήσης ε, των πυρηνικών όπλων. Εκεί που λέμε θέλουμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτές τις δύο, ε, αυτή την αλλαγή, ναι, αλλά αλλάζουν επί της ουσίας το νόημα. Συμφωνείτε με αυτή την προφορική τροπολογία. Ωραία, τότε επί του τμήματος 1 της 37 υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 37 πρώτο τμήμα, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Αυτό απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, αυτό εγκρίνεται. 39 του κύριου Βάιμερς. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ του κυρίου Παέτ. Κατά αποχές, ε, καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, να το δούμε. Μας λείπουν δύο. Θέλετε να ψηφίσετε. Ε, δεν πειράζει. Πέρας της ψηφοφορίας με μεγάλη πλειοψηφία. 44 του κυρίου Ντανζάν υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μικρή διαφορά όμως. Αιτιολογικές αναφορέ 1 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μια προφορική τροπολογία υπαριθμών 2, λέει ο μιλητή. υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 4, συντολογικές αναφορέ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Και περνάμε στην ε, συνολική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε σας παρακαλώ. It's closed. And uh, this has been adopted 61 to 1. Εγκρίνεται. 61 ψηφί υπέρ, 1 κατά. Εξαιρετική έκθεσή σας. Προφανώς κύριε Μίξερ, συγχαρητήρια. Αυτή ήταν ε, η ψηφοφορία για σήμερα. Συνεχίζουμε τη συνεδρία μας σε 5 λεπτά, οπότε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζωάου Βαλμέντα.